Πρόεδρε λέει όχι στην τροπολογία 1 και 2. Αντίθετα μπορεί να αποδεχτεί την τροπολογία 3 ε, του κυρίου Γκοζές. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι. Κύριε συνάδελφοι, εκ μέρους των Πρασίνων, ο Φιλίπ Λαμπέρτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ